Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Μάλστρομ, για τη συζήτηση αυτή, αγαπητοί συνάδελφοι. Αύριο η επόμενη σύνο... περίοδο συνόδου στις 8.30 το πρωί. Εύχομαι σε όλους καλό βράδυ.